για διορισμό του κυρίου Κέντ Ιόχανσον ως μέλος της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κροατία. Κοινή ε, κοινοβουλευτική, μειχτή μάλλον κοινοβουλευτική επιτροπή. Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι, οπότε το αίτημα αυτό εγκρίνεται. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας συζήτηση για την περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Η πρώτη συζήτηση για απόψε αφορά το Ιράν και τις τα πρόσφατα περιστατικά παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπέλντερ για δυόμιση λεπτά.